οι εργασίες της Επιτροπής μας. Αντί για τις τρεις, ε, όπως ε, γινόταν νωρίτερα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ε, μισή ώρα νωρίτερα. Όλες οι επιτροπές έχουν... Το κάνω αυτό σύμφωνα με απόφαση του Προεδρείου. Ε, σημεία 2 και 3. έγκριση των πρακτικών συνεδρία τη 7 η Σεπτεμβρίου. δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η δημόσια κρόση για την προστασία των δικαιωμάτων των εργατών σε προσωρινέ ε, ή επισφαλεί θέσει απασχόληση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στι 2.30. Και η κατάσταση έχει ω εξή. Πάνω από 60 εμπειρογνώμονε, πολλοί αναφέροντε και παρατηρητέ έχουν επιβεβαιώσει την προσέλευσή τους. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να συμμετάσχετε στην εκδήλωση αυτή. Κατόπιν δικού σας αιτήματο ε, θα, γίνει, θα πραγματοποιηθεί αυτή η ακρόαση. Και ήμασταν σε πολύ άσχημη θέση στην προηγούμενη μας ε, ακρόαση το εργαστήριο για τις αναπηρίες, ε, διότι την ώρα που ξεκίνησε η εκδήλωση εγώ και ένας βουλευτής ήμασταν παρόντες και καθ' όλη τη διάρκεια της ε, ακρόασης ε, δεν είχαμε ποτέ πάνω από δύο το πολύ τέσσερις ευρωβουλευτές. Σε μια χρυσή στιγμή είχαμε τέσσερις ευρωβουλευτές παρόντες. Αλλά κατά, κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της ε, ακρόασης συμμετείχαν μόνο δύο ευρωβουλευτές. Και αυτό δίνει πολύ κακή εικόνα θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μαγνητοσκοπούνται και μεταδίδονται σε όλη την Ευρώπη αυτέ οι ακροασει ε, και εμεί ε, λάβαμε απόφαση να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση. Εάν λοιπόν ε, ζητάτε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια εκδήλωση, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι θα είσαστε εσεί ή οι συνάδελφοί σα παρόντε. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στι 2.30 έχουμε 60 εμπειρογνώμονες παρατηρητές, πολλούς ανθρώπους παρόντες και παρακαλώ να βεβαιωθείτε ότι θα είσαστε και εσείς παρόντες. Δεν έχουμε κανένα σημείο στα διάφορα. Προχωράμε στην πρώτη ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε τοποθετήσει τις κάρτες σας στη συσκευή. Η πρώτη ψηφοφορία θα γίνει πάνω στην έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών. Ετήσια έκθεση της Επιτροπής μας για το έτος 2016. Ας προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία, εκτός αν ο εισηγητής θα ήθελε να πάρει το λόγο. Όχι? Ωραία. Προχωράμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Λυπάμαι, δεν βλέπω το όνομά σας. Ζαριανόπουλο. Και επί της διαδικασίας και επί της ουσίας να κάνω μια δήλωση για το θέμα το οποίο θα ψηφίσετε σε λίγο. Αφορά την απαλυφή, αφορά την, τροπολογία που έχουν καταθέσει οι πολιτικές ομάδες την απαλυφή μιας δραστηριότητας της Επιτροπής όσον αφορά την απόρριψη, το κλείσιμο της, Επιτρο... της αναφοράς σχετικά με τις γερμανικές αποζημιώσεις για τις ναζιστικές θηριωδίες κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα. Είναι αστήρικτη εντελώς νομικά με την έννοια ότι δεν παίρνει υπόψη της ούτε κάτι συμφωνίες για την ειρήνη του Παρισιού για τις πολεμικές αποζημιώσεις, δεν παίρνει υπόψη της παρά την αιτιολόγηση της ε, Κομισιόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεμβαίνει σε σχέσεις μεταξύ χωρών, παρεμβαίνει παντού στον κόσμο, το χαρακτηριστικότερο είναι ότι το σημαντικότερο σήμερα ζήτημα συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το Brexit και ποιο θα πληρώσει λιγότερα ή περισσότερα. Άρα είναι στην ευθύνη τη. Και τέλος είναι πολιτικά απαράδεκτη, διότι στην πραγματικότητα σιωπά δεν παίρνει θέση πάνω στα ναζιστικά εγκλήματα. Θα πρέπει ο καθένας να το σκεφτεί. Τη στιγμή που υπάρχουν πολιτικές ομάδες οι οποίες ζητάνε να στηθούν δίκες νηρευέργειες για τους κομμουνιστές, τι θα πει, τι σημαίνει η σιωπή για τα ναζιστικά εγκλήματα, Ποιο ωφελείται από αυτά. Θα πρέπει οι πολιτικές ομάδες να σεβαστούν τις ισίες του ελληνικού λαού και όλων των λαών κατά του ναζισμού και να πάρουν πίσω αυτή την τροπολογία είναι πραγματικά απαράδεκτη. Σε κάθε περίπτωση οι αγωνιστές της εθνικής αντίστασης και του δημοκρατικού στρατού στην Ελλάδα και το ΚΚΕ θα συνεχίσουν με ακόμα περισσότερη δύναμη για τη δικαίωση αυτού του αγώνα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μαριά, σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα να σας δώσω τώρα το λόγο. Ο κύριος Ζαριανόπουλος, ε, να σας πω ότι αυτή δεν είναι η στιγμή για ε, εσωτερική πολιτική συζήτηση ελληνικών θεμάτων. Αυτή είναι η στιγμή ψηφοφορίας. Να ψηφίσουμε, σας παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου, ο κύριος Ζαριανόπουλος. Listen. Ακούστε παρακαλώ, εάν ε, θεωρείτε, κύριε Ζαριανόπουλε, ότι εδώ μπορείτε να ορλιάζετε. Σας παρακαλώ όχι εδώ στην αίθουσα της Επιτροπής. Εγώ είμαι αρμόδια για την τάξη εδώ στην αίθουσα. Αν πραγματικά θέλετε να συζητήσετε, σας παρακαλώ εκτός αιθούσης, όχι εδώ. Εδώ ψηφίζουμε. Let's Προχωρούμε. Ο συζητητής πρέπει να μου δώσετε το λόγο. Όχι. I would like the floor as a rapporteur because... Θέλω το λόγο σε γιατί δώστε το λόγο και σε άλλα μέλη. Θα ήθελα λοιπόν το λόγο σε για ένα λεπτό. Please go ahead. Παρακαλώ. Go ahead. Θα είμαι πολύ σύντομα. Κύριε Πρόεδρε, καλούμαστε να εξετάσουμε την έκθεση. Νομίζω ότι από τις εργασίες που έγιναν και από τις ε, συζητήσεις με τους ε, Shadows έχουμε διαμορφώσει πάρα πολλές ε, τροπολογίες οι οποίες είναι σε επίπεδο συμβιβασμού, τα compromises και νομίζω ότι θα μπούμε στην ψηφοφορία. Μόνο στο σημείο 16 θέλω να αναφερθώ, στο οποίο ή στην έκθεσή μου εκφράζουμε τη λύπη μας ότι η αναφορά των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, υπαριθμών 22-14 του 14, σχετικά με τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις που οφείλονται προς την Ελλάδα, ενώ κρίθηκε παραδεκτή, I'm going to finish in one minute, κρίθηκε παραδεκτή το Σεπτέμβριο του 2015, δυστυχώς η πλειοψηφία των συντονιστών και όχι της Επιτροπής αποφάσισε να την κλείσει με τον ισχυρισμό ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι και λάθος και απαράδεκτο και πολιτικά επίσης λάθος και καλό τις ε, πολιτικές ομάδες οι οποίες έχουν καταθέσει τροπολογία επί της παραγράφου 16 του σημείου της έκθεσής μου που ζητούν να απορριφθεί αυτό το σημείο, να την αποσύρουν. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο πάνω στο οποίο υπάρχει συζήτηση και διαφωνία. Και τις καλώ λοιπόν να αναλογιστούν τις ιστορικές τους ευθύνες και να αποσύρουν την τροπολογία αυτή με την οποία ζητούν να απορριφθεί η παράγραφος 16 της ε, εκθέσεώς μου. Επιμένω σε αυτό, αυτή είναι η θέση που έχω ως εισηγητής, δικαιούμαι να το πω, ε, με βάση και τη συζήτηση που διεξήχθη και μπορούμε, να, προχωρήσουμε στην, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία αφού κάνω την έκκληση στις πολιτικές ομάδες να αποσύρουν τη δικιά τους τροπολογία και να παραμείνει σε ισχύ η παράγραφος 16 της εκθέσεώς μου για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Σας ευχαριστώ. Listen, now I think that we need... Ακούστε, θα πρέπει να είμαστε όλοι λογικοί. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Παραγραφός 1, τροπολογία 43, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, να ελέγξουμε, να επαληθεύσουμε παρακαλώ. There is one Okay, is the vote finished? I think it is. Yes. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Τροπολογία 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Είναι πολύ μικρή η διαφορά. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ωραία. 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Παρακαλώ. And the vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται κατά τρεις ψήφους. 67 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Συμβαστική 1. Παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 69 το πρώτο τμήμα υπέρ. Όχι λάθος, 72 διορθώνει η πρόεδρος. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 78 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Παρακαλώ. And the vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές. ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 έως 111 ταυτόσημες είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. And we close the votes, vote, and it is... Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. 112. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται κατά τρεις ψήφους. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 Θέλετε η ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 5. Άρχεται η ψηφοφορία. It is rejected. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ε, να μ' ακούτε. <laughs> Θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα έτσι. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά, κατά αποχές απορρίπτεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Ποια θέλετε να επαληθεύσουμε, 21. Άρχεται η ψηφοφορία για την 21, ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά αποχές να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν είμαι και ποτέ σίγουρη, ποτέ δεν έχουμε την ίδια πλειοψηφία. Εγκρίνεται κατά δύο ψήφους. Έχουμε μία προφορική τροπολογία. Η προφορική αυτή τροπολογία αφορά την αιτιολογική σκέψη J λέει ενώ αρκετά μεγάλος αριθμός αναφορών συζητώνται δημόσια στις ε, ε, συνεδριάσεις της Επιτροπής ε, και οι αναφέροντες έχουν δυνατότητα συμμετοχής συμβάλλοντας ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής. Το 2016, 201 αναφέροντες ήταν παρόντες, ενώ 61 συμμετείχαν παίρνοντας το λόγο στις συζητήσεις της Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ήταν παρόντες 201 ε, αναφέροντες, αλλά δεν πήραν όλοι το λόγο. Μπορούμε παρακαλώ να ε, ψηφίσουμε αυτήν την τεχνική ε, τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. 37. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά ε, η ηλεκτρονική επαλήθευση 42 λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται τελική ψηφοφορία πάνω στο σχέδιο γνωμοδότησης στο σύνολό του. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κύριε Πρέντα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Παίρνω το λόγο για να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τον κανονισμό. Μια μεγάλη πλειοψηφία, 19 υπέρ 9 κατά, είχαμε, αποφασίσαμε να διαγράψουμε την παράγραφο 16. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε από αυτή την έννοια να διαγράψουμε και το, αντίστοιχο εδάφιο ε, της ιδιαιτιολογικής έκθεσης. Πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε επί τη βάση του κανόνος 52α που αναφέρει τα εξής. Η παράγραφος 2 ε, του κανόνα αυτού λέει η, τελική έκθεση είναι ευθύνη του εισηγητή και δεν θα τίθεται σε ψηφοφορία. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να συνάδει με το κείμενο του, ε, της έκθεσης ε, όπως ψηφίστηκε, καθώς επίσης και με τις τροπολογίες που έγιναν δεκτές. Ο πρόεδρος μπορεί να διαγράψει κομμάτια της αιτιολογικής έκθεσης. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος, και ευχαριστώ πολύ που το θέτε υπόψη μας. Κύριε Μαριά, εσείς δέχεστε να υιοθετηθεί το κείμενο σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Πρέντα. Ε, ή την απόφαση θα πάρω εγώ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες βγάζουν αλλεργία όταν ακούν για την διεκδίκηση εκ μέρους της Ελλάδος των γερμανικών αποζημιώσεων. Ένα θέμα που έχει καθοριστεί με απόφαση της Συνθήκης Ειρήνης του 1946. Μια διεθνής απόφαση η οποία ισχύει. Επομένως, ό,τι και αν ψηφιστεί νομικά εδώ δεν έχει καμία αξία, διότι το διεθνές δίκαιο υπάρχει, οι διεκδικήσεις της Ελλάδος ισχύουν και δεν διαγράφονται και να είστε βέβαιος κύριε Πρέντα και οι υπόλοιποι ότι αυτό θα γίνει αποδεκτό και θα υπάρξει η πλήρης δικαίωση των θυμάτων του ναζισμού, οι οποίοι ζητούν πλήρη αποκατάσταση και οι πολεμικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο και οι αποζημιώσεις των συγγενών των θυμάτων. Επομένως εδώ η μικροπολιτική την οποία κάνετε δεν πρόκειται να περάσει. Αυτό ε, προς το πολιτικό μέρος. Πήρατε την απόφαση για την τροπολογία 16 για να ανατρέψετε την ε, ρύθμιση που υπήρχε μέσα στην έκθεσή μου. Και εγώ, παρότι εισηγητής, καταψήφισα την έκθεση τελικά, στο τέλος. Διότι για μένα κυρίαρχο θέμα είναι ότι σε αυτήν εδώ την Επιτροπή έχετε κάνει κάθε προσπάθεια να απορρίψετε κάθε προσπάθεια και κάθε αναφορά στις γερμανικές αποζημιώσεις. Και είναι δύο οι δράσεις που έγιναν εδώ. Πρώτον, επί τρία χρόνια συνεχώς ως Επιτροπή απορρίπτεται την πρότασή μου για δημόσια ακρόαση και συζήτηση για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Δεν τολμάτε καν να συζητήσετε δημόσια το θέμα αυτό. Αν είχατε δίκιο γιατί άραγε δεν θέλετε να συζητηθεί. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, μέσα στην Επιτροπή, μέσα στους συντονιστές, ενώ κρίθηκε η αναφορά 22-14 του 14 των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος ως παραδεκτή, φτάσατε στο τέλος να πείτε ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων. Επομένως, καταλάβετε το, ότι με μαγικά τρίκ δεν μπορείτε να διαγράψετε την ιστορία. Έρχομαι λοιπόν ως προς τον ισχυρισμό του κυρίου Πρέντα. Ως προς τον ισχυρισμό του κυρίου Πρέντα. I will continue. I will continue. This, this committee is getting unmanageable with you taking... Αυτή, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την επιτροπή αν παίρνετε το λόγο και δεν τον δίνετε. Μου δώσατε το λόγο και πρέπει να απαντήσω στις προτάσεις του κύριου Πρέντα. Είμαι ο εισηγητής. εάν διαβάσετε το σημείο 2, τι λέει. Πρώτα απ' όλα, ουδέποτε σε αυτή την επιτροπή και σε καμία άλλη επιτροπή δεν αλλάξατε το explanatory statement του εισηγητή. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό κύριε Πρέντα. και αυτά που ζητάτε είναι απίθανα. Δεύτερον, Δεύτερον. Mr. Δεύτερον. No. Δεύτερον. I, I will finish my Mr. arguments. Mr. I will finish Can... my arguments. Listen, I happen to be the chair of this. Πάρε λίγο τα αγγλικά γιατί δεν μπορώ να... Κύριε Πρέντ, ε, Μαριά σας παρακαλώ, δεν με αφήνετε να τελειώσω και να εκφράσω τα επιχειρήματά μου. Θέσατε μία ερώτηση προς εμένα και θα απαντήσω την ερώτησή σας. Ναι, θα απαντήσω στην ερώτησή σας πρέπει να καταλάβετε ότι εδώ πρόκειται για Δημοκρατική Επιτροπή και δεν είναι μια επιτροπή η οποία είναι ε, βάση του τι επιθυμείτε και νομίζετε εσείς. Έχω το λόγο λοιπόν και θα συνεχίσω και σας παρακαλώ μετρήστε, δώστε μου χρόνο να ε, απαντήσω. Απαντά σε σχόλιο εκτός μικροφώνου ο κύριος Μαριάς. Λέει, λέει το σημείο 2 It falls, to the chair, it falls to the chair of the committee to delete the explanatory statement. Επομένως, πρέπει πρώτα διαδικαστικά να πάρετε την έκθεση όπως διαμορφώθηκε μετά την ψηφοφορία. Πρέπει να την αποτυπώσετε, πρέπει να τη διαβάσετε και αφού τη διαβάσετε να δείτε αν υπάρχει το explanatory statement και αν αυτό έχει σχέση. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να πάρετε απόφαση. Δεύτερον, αυτό το οποίο αναφέρουμε στο explanatory statement αφορά, αφορά τη γνώμη του εισηγητή. Επομένως, θα πρέπει να παραμείνουν τα σημεία αυτά. Κάθε άλλη απόφαση η οποία θα ληφθεί είναι αντιδημοκρατική. Listen, Κοιτάξτε, δεν έχω καμία δυνατότητα εδώ στην επιστροφή να σας ε, κόψω το μικρόφωνο. Αν είχα αυτή τη δυνατότητα θα σας το είχα κλείσει το μικρόφωνο. Εσείς μου δώσατε το λόγο και θα πρέπει να μου δώσετε χρόνο. Δεν μου βάλατε κάποιο χρονικό όριο και επομένως μπορείτε να μου βάλετε όπως επιθυμείτε. Κύριε Μαριά, σας έδωσα το λόγο, αλλά περίμενα να τον επιστρέψετε κιόλας βάσει του άρθρου 52α παράγραφος 2 του κανονισμού εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής μπορώ να διαγράψω το επεξηγηματικό ε, σημείωμα πλήρως ή εν μέρη. Και εγώ έχω πρόθεση να διαγράψω την παράγραφο για τις αναφορές που αφορούν τις συνέπειες ε, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που περιλαμβάνονται εκεί. Και αυτό γίνεται ακριβώς βάση του κανονισμού και αυτό ακριβώς κάνω αυτή τη στιγμή. Απλώς διαδικαστικά. Θέλω να επαναλάβετε τι διαγράψατε από, την, από, την, από το explanatory statement. Ακριβώς για τα πρακτικά. Τι διαγράψατε. Διαβάστε ακριβώς τι διαγράψατε για τα πρακτικά. Διαγράφω την τελευταία παράγραφο για το θέμα αναφορές που αφορούν ε, τα θέματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η παράγραφος διαγράφεται από εξεγερματικό σημείωμα. Αυτή είναι η μόνη παράγραφος που διαγράφεται. Ναι, αυτή είναι η παράγραφος που διαγράφω. Και την απόφασή σας μετά. Now, I am very sorry for, for this. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την πολύ δυσάρεστη ατμόσφαιρα εδώ στην ε, ε, Επιτροπή. Εσείς φταίτε κύριε Μαριά. Και ζητώ συγγνώμη εκ μέρου σα τώρα, διότι από ό,τι κατάλαβα εσεί δεν θα ε, ζητήσετε ποτέ συγγνώμη. Ως πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής ζητώ συγγνώμη στου συναδέλφου εκ μέρου σα για τη συμπεριφορά σας. Ε, η συμπεριφορά μου ήταν άριστη. Ήταν άριστη. Από εκεί και πέρα να κρατήσετε πρακτικά για το τι διαγράψατε ακριβώς. Έχει μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ πολύ. Now, let's, let's proceed Τώρα, να περάσουμε στη δεύτερη ψηφοφορία για την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. κυρία Τούμ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω να διαγράψετε από τη συμβαστική πρόταση J την πρόταση 157, ε, διότι αυτό το οποίο αναφέρεται σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό το σκεπτικό της πρότασής μου και επίσης θα ήθελα να αποσύρετε την 157 ε, από τον κατάλογο ψηφοφοριών. Ευχαριστώ πολύ. Did I understand you correctly? You wanted... Αν κατάλαβα καλά, θέλετε να εξαιρεθεί από το συμβιβασμό και να... αλλά να ψηφιστεί... Α, όχι και από τα δύο. Ωραία. Αποσύρετε λοιπόν πλήρως την ε, τροπολογία σας. Ωραία, το σημειώνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 78, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 81, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Επαλήθευση για την 84. Υπάρχει ένας επιπλέον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 Οι φιλελεύθεροι πρέπει να είναι τρει, τρει είμαστε και οι σοσιαλιστέ είναι οχτώ. Εσεί δεν ψηφίζετε, εντάξει. Έχετε βάλει την κάρτα σα, Όχι από ό,τι φαίνεται. Μπορεί να έκανα και λάθος το μηχάνημα. Ας ξαναψηφίσουμε. 30 κάρτες έχουμε. Η Γκουε, πόσες ψήφους έχετε, δύο. Το ECR είναι δύο. Η SND είναι 8. Κάποιος πρέπει να έχει ξεχάσει την κάρτα του στο μηχάνημα και να έφυγε. Βλέπετε κάποια κενή θέση με κάρτα στο μηχάνημα. Κάποιο Κάποιος έχει προσθέσει μια κάρτα στο μηχάνημα, αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι. Μπορούμε να σταματήσουμε στις 29 ψήφους. Χρειάζομαι τρεις ακόμα ψήφους. Ναι, παρακαλώ όλοι αφαιρέστε τις κάρτες σας. Και τώρα για να δούμε, υπάρχει μία κάρτα κάπου. Σας παρακαλώ σταματήστε, κάποια υπάρχει μία κάρτα. Η κυρία Αλμπιόλ μπορεί να βγάλει την κάρτα της. Και η κυρία Άντερσον επίσης. Κύριε Κοτσολίνο, μπορείτε να βγάλετε την κάρτα σας. Εντάξει, τώρα είναι κενό. Να προσθέσουν τις κάρτες τους οι σοσιαλιστές. Είμαστε 8. Εντάξει, οι σοσιαλιστές είναι 8. Το ΕΛΚ τώρα. Η πράσινη τώρα. Okay. Now, the GUE. Η Γκουε, e. τρεις ψήφους επίσης. Okay. ECR. Το ECR, τις δύο κάρτες τους. And Alde would put in the three. Και η φιλελεύθερη τρεις. Και το EFTD, μία το enf 1 και λογικά είμαστε τάξη. Για να ψηφίσουμε λοιπόν που ήμασταν. Ε, γινόταν επαλήθευση της συμβαστικής τροπολογίας 84. Επαλήθευση της τροπολογίας 84. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία D υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, πρέπει να κάνουμε επαλήθευση και εδώ. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 93 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση και σε αυτό. εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ή e, υπέρ. Θέλετε παλήθευση της 96. Άρχεται η ψηφοφορία για την 96. Πέρας της ψηφοφορίας ε, απορρίπτεται. βασική τροπολογία ή, e, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 102, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Α, όχι, καταπίπτει. Δεν ψηφίζουμε. Έχετε δίκιο. Τροπολογία 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμ... βασική τροπολογία H, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 120. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 122, υπέρ, Κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία I υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 123 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 129 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία... Ε, α, πίπτη, συγγνώμη. 127 υπέρ. Κατά αποχές ε, πρέπει να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για έλεγχο στην 127. Εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 133 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ, κατά, α, πρέπει να επαληθεύσουμε, άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας, εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 135 υπέρ κατά αποχές πρέπει να επαληθέσουμε και αυτήν. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 133 εγκρίθηκε, πάμε στην 139 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά αποχές πρέπει να επαληθεύσουμε. Ακόμα είναι ανοιχτή ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. «147 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται». «155 υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για έλεγχο για την 155. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Βλέπετε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελέγχονται. Συμβαστική τροπολογία K υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 190 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 194 έχει αποσυρθεί. 163. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. The vote is open and closed. Απορρίπτεται. 165 υπέρ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 165 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και πάλι επαλήθευση. Έναξη ψηφοφορίας. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση και εδώ. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική L. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 167. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση. Αν σηκώνετε το χέρι σας δεν χρειάζεται να επαληθεύουμε συχνά αλλά λίγη σοφορία εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και πάλι βαλθεύουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται με διαφορά τριών ψήφων. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση N. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία O. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 189. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 188. Έχει αποσυρθεί 188. 191. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Look at that. That was closed. That is now closed. Ωραία, απορρίφθηκε. 192, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλληλεκτρονική επαλήθευση. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 193 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε παράγραφος 2 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε παράγραφος 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. And vote. It has been adopted by one. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Okay, maybe we should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 Αποχές. Εγκρίνεται. 200 έχει αποσυρθεί. 201 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ελεκτρονική επαλήθευση. Απορρίπτεται. Ισοψηφία απορρίπτεται. Ε, τελική εκτισή, το προλογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 ε, καταπίπτει, 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 5. Όλα θα εγκριθούν, μου φαίνεται. Θέλετε να τα ομαδοποιήσουμε όλα μέχρι την τροπολογία 17. Μέχρι τη 17. Όλα μαζί. Όχι, όχι, όχι αρνούνται. Γκουε δεν θέλει. Και το FTD δεν θέλει. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, Εποχέ. εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, Εποχέ. απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, Εποχέ. εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, Εποχέ. εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, Εποχέ. εγκρίνεται. 32 υπέρ, Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα. And it Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. ...37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 43 πρώτο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 επαλήθευση για τη 49 επαλήθευση τη 49 απορρίπτεται «45 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται». 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική πρόταση π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική επαλήθευση για την 59 εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το σύνολο του κειμένου. Τελική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. This was a very tight... Πολύ δύσκολη ψηφοφορία. Ας προχωρήσουμε τώρα στην κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 1. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω πρέπει να επαληθεύσουμε.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 αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έχουμε εδώ μια χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα της χωριστής ψηφοφορίας, ε, τροπολογία 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 καταπίπτει.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 την αποστολή στην Ισπανία. It's a very complicated item. Let's go to Amendment 1, the first part. Τροπολογία 1. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επαλήθευση. The vote is open. And it is closed and adopted. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Καταπίπτει, συγγνώμη. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά πάμε στην τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 23. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 19. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται με μία ψήφο. Όλα στον πόντο κρίνονται σήμερα. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Καταπίπτει. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9, όχι, την 55 πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, 58, το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αυτό πρέπει να το επαληθεύσουμε. 68 επαλήθευση. Απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, πρέπει να επαληθεύσουμε. 71 Άρχεται η ψηφοφορία τώρα για έλεγχο.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 Μικρόφωνο παρακαλώ. Θα μπορούσαμε να επαληθεύσουμε την τροπολογία 70, γιατί νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τροπολογία 70. Έχει εγκριθεί. Α, εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να περάσουμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Να δώσω το λόγο στην κυρία Πιτέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρέμβω για τις διάφορες ψηφοφορίες εξ ονόματος ε, του ΕΛΚ. Καταρχάς, ε, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο το έχουμε εδώ και δεκαετίες και αφορά τις κυβερνήσεις ε, της Ισπανίας οι οποίες ε, ήταν είτε της δεξιάς είτε της αριστεράς. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο ε, απασχολεί ιδιαίτερα την κοινωνία και αποτελεί και αντικείμενο συζητήσεων και πρέπει να έχουμε μια αντικειμενική γνωμοδότηση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τα διάφορα στοιχεία και ε, τα έγγραφα, αλλά δεν υπάρχει μια πλήρης αξιολόγηση της κατάστασης. Για παράδειγμα, η βάση δεδομένων στοιχείων DNA, η οποία θα πρέπει να καταρτιστεί. Σε κάποιες περιπτώσεις δίνεται εντύπωση ότι η Ισπανική κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς ε, θέλαμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη δήλωση. Ευχαριστώ πολύ. E Ευχαριστώ πολύ. Το ΕΛΚ θα ζητήσει λοιπόν και μια γνωμοδότηση μειοψηφία ε, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 4 του κανονισμού και αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε ε, μια γραπτή δήλωση η οποία δεν θα υπερβαίνει σε 100 λέξεις και έχετε προθεσμία μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης. Ε, ωραία. Αυτό θα γίνει και θα προχωρήσουμε τώρα και να καλωσορίσω την Ένωση Λασκέλης για την κατάσταση της, της απασχόλησης ε, των καμαριέρων ξενοδοχείων στην Ισπανία. Να ζητήσω από τους συναδέλφους που δεν σκοπεύουν να συμμετέχουν στη συζήτηση, σας παρακαλώ να αποχωρήσετε ησύχως όσο το δυνατόν. 9. Ωραία λοιπόν, ε, η αναφορά 99 είναι αυτή τη στιγμή στην ημερήσια διάταξη και να δώσω το λόγο στην αναφέρουσα για να λάβει το λόγο για 5 λεπτά. Το πολύ. Άγχελες Μουνιώθ Ροντρίγες, έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Ε, είμαστε η Ένωση Λασκέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχετε το αίτημά μας εξ ονόματος όλων των γυναικών που εργάζονται ως καμαριέρες στην Ισπανία. Γνωρίζουμε τι ευθύνη προϋποθέτει να συζητούμε για την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια, διότι πρόκειται για έννοιες οι οποίες είναι εγγενεί των ανθρώπων σε όλες τις συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς καμία εξαίρεξη και φυσικά βρισκόμαστε εδώ διότι πάρα πολλοί παράγοντες δεν μας επιτρέπουν να απολαμβάνουμε αυτών των δικαιωμάτων στην άσκηση της καθημερινής μας δουλειάς. Στο τμήμα των διαμερισμάτων στο οποίο ανήκουμε ε, ασχολείται με την ε, ε, ευημερία και την άνεση των πελατών των ξενοδοχείων και η κατηγορία μας είναι καμαριέρα ξενοδοχείου και πρέπει να διατηρούμε καθαρά και να εγγυόμαστε την καθαριότητα σε κοινόχρηστους χώρους και σε δωμάτια ξενοδοχείων. Πρόκειται για μια ε, φυσική δουλειά, πολύ σκληρή ε, και ε, κανείς δεν θέλει να μένει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου που να μην είναι καθαρό. Είμαστε το 30% του πρωτοσωπικού των ξενοδοχείων και είμαστε περίπου 100.000 καμαριέρες και υπάρχουν ε, αυτή τη στιγμή ε, χιλιάδες γυναίκες ε, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζονται με αυτές τις συνθήκες. Οι κυβερνώντες το αποκαλούν αυτό οικονομική ανάπακαμψη. Οικονομική ανάκαμψη. Είμαστε το 30% των, του προσωπικού των ξενοδοχείων δεν είμαστε αριθμοί, παρά το γεγονός ότι είμαστε περίπου 100.000 καμαριέρες σε όλη τη χώρα και τα, ε, ποσά, το η αριθμή των επισκεπτών είναι 84 εκατομμύρια, 12% ε, αύξηση κάθε χρόνο και τα οικονομικά ωφέλη αποτελούν περίπου το 16% του ΑΕΠ. Και αυτά ε, φυσικά ε, κυμαίνονται συνεχώς ε, και φυσικά θα πρέπει και εμείς να σας δείξουμε εδώ τι γίνεται με αυτές τις διακυμένσεις. Καταρχάς υπάρχουν ασθένειες οι οποίες δεν αναγνωρίζονται γνωρίζονται ως επαγγελματικές ασθένειες λόγω της δουλειάς μας. Το 90% έχουμε κάποια προβλήματα στο ομοιοσκελετικό σύστημα. Το 71% παίρνει φάρμακα καθημερινά για να δείξει τους πόνους και την επιβάρυνση της εργασίας. Το 96% πάθει από άγχος ε, λόγω του πόνου και της πίεσης. Το 28,45% έχει συμπτώματα βαριάς κατάθλιψης και το 17% ήπιας κατάθλιψης. Ε, και μπορεί να ακούγεται επίπονο και μόνο να τα ακούτε, αλλά αν θέλετε να δείτε πραγματικά μια επίπονη κατάσταση, μπορείτε να δείτε τα χέρια της ε, ε, συναδέλφου εδώ που μας συνοδεύει. Είναι φρενήρηση η ρυθμή και πρέπει να Καθαρίζουμε περίπου 400 δωμάτια το μήνα, περίπου κατά μέσο όρο δηλαδή 40 δωμάτια την ημέρα και 20 μπάνια και έχουμε χιλιά, ε, πολλά κιλά που πρέπει να σηκώνουμε, χρησιμοποιούμε χημικά προϊόντα και κάνουμε περίπου 11.000 βήματα, περίπου 11 με 12 χιλιόμετρα σε φρενήρις ρυθμούς, χωρίς χρόνο να φάμε, για να πάρουμε 800 ευρώ μειχτά, ε, ανάλογα με τη σύμβαση που έχουμε έχουμε έρθει εδώ στις Βρυξέλλες γιατί μπορούμε να αποφύγουμε τις ασθένειες που, λαμβα... παθαίνουμε από την εργασία. Εάν τηρούνταν η νομοθεσία δεν θα βρισκόμασταν εμείς εδώ. Εφαρμόζοντας την νομοθεσία ε, και ούτε καν τα ασφαλιστικά ταμεία δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία. Θα πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία για την ε, πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και να αγκιάται και η συμμετοχή των εργαζομένων σε όλη τη διαδικασία. Ε, Επίση, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στου ηθήνοντε ότι πρέπει να τηρηθεί νομοθεσία και να τιμωρηθούν αυτοί που δεν την τηρούν, όπω καθορίζεται από το άρθρο 40, σημείο 2 του Ισπανικού Συντάγματος. Πέρα από το γεγονό ότι γίνεται εξωτερική ανάθεση για τι υπηρεσίε, ε, που σημαίνει ότι μείωθηκαν οι μισθοί μα κατά 40% και καταργήθηκαν κάποια θεμελιώδη δικαιώματα, ε, ε, φτωχοποίηση των γυναικών, επισφάλεια, απάτη στι συμβάσει, υπερφόρτωση τη εργασία και υπερβολική προσπάθεια που επιδεινώνουν την κατάσταση τη υγεία μα και την ποιότητα τη ζωή μα. Καταγγέλνουμε επίσης και την κατάσταση πολλών εργαζομένων γυναικών με αναγνωρισμένες αναπηρίες μέσω προγραμμάτων ένταξης και ειδικής απασχόλησης με επιδοτήσεις από δημόσια κονδύλια και από ευρωπαϊκά κονδύλια. Κάποιε επιχειρήσει κερδοσκοπούν με κάποιε συγκεκριμένες κατηγορίες ε, ε, και καταχρώνται αυτές τι ε, συγκεκριμένε συνθήκε. Ε, και πραγματικά υπάρχουν συγκεκριμένες νομοθεσίες που αφορούν χώρους εργασίας ε, και επιβάρυνση της εργασίας, ε, κοινωνικο-οικονομικούς κινδύνους και γι' αυτό ακριβώς ζητούμε μελέτη από μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα κάνει πραγματική πραγματογνωμοσύνη των συνθήκων εργασίας μας, διότι η υγεία δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλες σας που ήρθατε εδώ και σας ευχαριστούμε πολύ που η μία στηρίζεται την άλλη. Δεν είναι κάτι απλό αυτές τις μέρες. Πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο ε, και να δρούμε ενωμένοι. Κυρία Αλμπιόλ, το λόγο. I, Συγγνώμη, έκανα ένα μεγάλο λάθος πρέπει να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Κομισιόν, στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, Γιάνν Βίλεμ Έμπελινγκ, από το τμήμα, ε, από τη μονάδα απασχόληση. Ονομάζομαι Έμπελινγκ, εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση ΕΜΠΛ, στην, στο τμήμα ασφάλειας και υγείας. Ε, Η, ε, το σωματείο Λασκέλης έχει πάνω από 2.000 μέλη στην Ισπανία και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενθαρρύνουν τις Ισπανικές αρχές ε, να μεριμνήσουν έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τις ε, ευρωπαϊκές οδηγίες αφενός και την εθνική νομοθεσία αφετέρου. για να βελτιωθεί η κατάσταση. Η Κομισιόν προετοίμασε κάποιες γραπτές παρατηρήσεις, ε, θα σας τις ε, συνοψίσω. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ε, νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά τα θέματα προβλέπει η πρόεδρο αυτά κείμενα ότι οι εργοδότες θα πρέπει να εξετάζουν και να αξιολογούν τους ενδεχόμενου κινδύνους και να παίρνουν και τα κατάλληλα μέτρα. Για παράδειγμα, αν οι εργαζόμενοι πρέπει να σηκώσουν μεγάλα βάρη. Θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να εγκαθίστανται μηχανήματα που να βοηθούν του εργαζόμενου. Επίση, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να επιθεωρούν ε, τα, τους χώρους εργασίας, ε, και να παρακολουθούν τα μέτρα που λαμβάνονται. Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να μεταγραφούν από τα κράτη-μέλη, αλλά τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή τους ε, και για τις επιθεωρήσεις ε, και για την επιβολή κυρώσεων. Να προσθέσω ότι από πλευράς Κομισιόν έχει εκδοθεί μια ανακοίνωση φέτος 2017 ε, και κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για τον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας ασφάλειας και υγείας και της πολιτικής ασφάλειας και υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γίνεται ένας απολογισμός ε, των, της νομοθεσίας των τελευταίων ετών και αναφέρεται ότι έχουν έχει επιτευχθεί πρόοδος αλλά εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά προβλήματα, μειοσκελετικές διαταραχές, για παράδειγμα, είναι ένα από τα προβλήματα οποία αναφέρονται πολύ συχνά και που καλύπτονται από ευρωπαϊκές οδηγίες. Τώρα έχουμε και τις κατευθύνες γραμμές, οι οποίες απευθύνονται κυρίως στους εργοδότες με συγκεκριμένες ε, συμβουλές για το πώς πρέπει οι εργοδότες να λαμβάνουν μέτρα για να αποφεύγονται τέτοιου είδου μειοσκελετικές διαταραχές. Έχουμε, έχουν διοργανωθεί και εκστρατείες πληροφόρησης ε, ε, και από την ε, Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της χωροασίας και από το, την Επιτροπή ΣΛΙΚ των Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας και γενικότερα τα κράτη-μέλη συνεργάζονται για να ε, ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές ε, και να εξετάζουν κάθε φορά το πώς μπορούν να βελτιώσουν τις επιθεωρήσεις και την ε, συμμόρφωση επιτόπου. Αυτά προς το παρόν. Thank you very much for... ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος του συνάδελφου. Κύριε Αλμπιόλο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τις αναφέρουσες ε, και να υπογραμμίσω την αξία του αγώνα των Λασκέλης. Είναι ένας σύλλογος που απαρτίζεται κατά βάση από γυναίκες οι οποίες ε, χαρακτηρίζονται από επισφάλεια στην εργασία, με... εργάζονται υπό την απειλή της απόλυσης. Παρόλα αυτά κατάφεραν να συνδικαλιστούν, να να οργανωθούν και ε, οι διεκδικήσεις τους φτάνουν όχι μόνο παντού στην Ισπανία αλλά μέχρι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, συγχαρώ για αυτό τον αγώνα σας. Και το γεγονό ότι βρίσκονται εδώ σήμερα, το γεγονό ότι έχουν υποβάλει αυτή την αναφορά, οφείλεται στο ότι το κράτο στην Ισπανία δεν αναλαμβάνει δράση έτσι ώστε να θέσει τέλο σε αυτή την κατάσταση εκμετάλλευση και επισφάλεια την οποία μα παρουσίασαν χιλιάδες ε, γυναίκες ε, είναι θύματα αυτής της κατάστασης στην Ισπανία. Εμείς έχουμε ευθύνη ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, διότι υφίστανται ευρωπαϊκές οδηγίες, για παράδειγμα της ασφάλισης και της υγείας στο που δεν τηρούνται. Ε, το, υπάρχει οδηγία για τον συνδυασμό της προσωπικής με, ε, με την επαγγελματική ζωή, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Χάρτα, ε, υπάρχουν τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία καταπατούνται. Συνεπώς θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση που να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Προφανώς το Ισπανικό κράτος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις οδηγίες. Όταν όμως ένα κράτος δεν εφαρμόζει κάποιες οδηγίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ανοίξει τα χέρια της και να πει ότι είναι θέμα του κράτους. Αν το κράτος δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε να τις εφαρμόσει ε, και ενδεχομένως να ανοίξει διαδικασίες επί παραβάση η Ευρώπη έχει ε, ευθύνη διότι η Ευρώπη έχει πολύ συχνά ε, αναλάβει πρωτοβουλίες για εργασιακές μεταρρυθμίσεις πολύ συχνά βάναυσες που οδηγούν σε τέτοια κατάσταση αυτές και άλλες γυναίκες. Ε, έχουν χειροτερέψει οι μισθοί, έχουν μειωθεί οι μισθοί, έχουν χειροτερέψει οι συνθήκες εργασίας στο πλαίσιο αυτών των εργασιακών μεταρρυθμίσεων. Η εταιρείε αυτές ε, οι οποίες ε, αναλαμβάνουν την ανάθεση αυτή δίνουν υπεργολαβία αυτές τις αναθέσεις σε άλλες εταιρείε οι οποίες πραγματικά δρούν ε, χωρίς έλεγχο, ανεξέλεγκτα. Το προσωπικό χάνει δικαιώματα, οι κοπέλες εδώ μίλησαν για τους χαμηλούς μισθούς, για τα μεγάλα βάρη τα οποία ε, σηκώνουν για την κατάσταση των εργαζομένων με αναπηρίες, για ασθένειες οι οποίες δεν αναγνωρίζονται. Χρειάζεται απάντηση. Τελειώνω προτείνοντας τα εξής. Ε, προφανώς αυτό που προτείνουν οι ίδιες οι, οι αναφέρουσες να εξεταστούν οι συνθήκες εργασίας τους, αλλά ως Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να κάνουμε ένα ακόμα βήμα. Και είναι μια ευκαιρία Ενδεχομένω να υποβάλουμε μια, ένα προφορικό ερώτημα προς την Κομισιόν για τις συνέπειες των ε, εργατικών μεταρρυθμίσεων των, και τη ε, επισφάλεια στην εργασία. Γιατί ε, υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο η Κέλλης. Έχουμε τους εργαζόμενους στα οι υπάλληλοι σε κάποιες χώρες, οι δημόσιοι υπάλληλοι σε κάποιες χώρες. Συνεπώς η, μια προφορική ερώτηση στην Κομισιόν για την ε, επισφάλεια και βέβαια να ε, αντιχύσει μέσω ημών η κατάσταση αυτών των ε, καμαριέρων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, πληροφοριακά, να σας πω τα εξής ασφαλώς και μπορούμε ως Επιτροπή να πάρουμε πολλά μέτρα, αλλά να υποβάλουμε προφορική ερώτηση στην Κομισιόν είναι μια απόφαση η οποία λαμβάνεται από τους συντονιστές. Οπότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στον συντονιστή σας Έτσι δρούν οι πολιτικέ ομάδε. Δεν μπορούμε να πάρουμε μια τέτοια απόφαση εμεί εδώ σήμερα, περί προφορική ερώτηση. Άλλα μέτρα μπορούμε να λάβουμε, θα το δούμε αργότερα. Κυρία Γκαρθία Πέρες. Καλώ ήρθατε. Για πρώτη φορά είστε εδώ, νομίζω, έτσι δεν είναι. Δεν σα έχω ξαναδεί. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω ε, την, το Σωματείο Λασκέλης που εκπροσωπεί τις ε, καμαριές ξενοδοχείων. Τη συγχαίρω για τα αιτήματά τους, για τις διεκδικήσεις τους, για το ότι θέτουν προς συζήτηση ένα ολόκληρο αγώνα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των καμαριέρων ξενοδοχείων. Τις γνωρίζουμε, έχουν διοργανώσει και ίδιες και άλλα συνδικαλιστικά όργανα και πλατφόρμες μια ολόκληρη εκστρατεία ενημέρωσης. Ε, συμμεριζόμαστε τα αιτήματά τους και δίνουμε συνέχεια σε, πολιτικό, σε πολιτική συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. οι συνέπειε της εργασιακή ε, ε, των εργατικών μεταρρυθμίσεων στην Ισπανία οδήγησαν στην αύξηση της επισφάλειας στην Ασία. Τα, ε, οι συμβάσει εργασία είναι συμβάσει φτώχεια. υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ισπανία μια ολόκληρη, ένα τμήμα του εργατικού πληθυσμού που ζει κάτω από το κατόφλι της φτώχειας και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και τις πιο βασικές του καθημερινές ανάγκες. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να αντιληφθεί αυτήν την κατάσταση. Επίσης γίνεται λόγος για, την, για το ότι η φτώχεια γίνεται όλο και πιο θηλυκού φύλου. Η ε, έξοδος από την οικονομική κρίση σε πολλές ε, χώρες ε, ε, ερμηνεύεται μόνο ως βελτίωση των μακροοικονομικών στοιχείων, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την πραγματική κατάσταση των ανθρώπων ε, με τις μεγάλες σημαντικότατες ε, διαφορές ε, που υφίστανται σε πλούτο, σε εισόδημα και σε συνθήκες εργασίας. Οι, ξενο... οι καμαριές ξενοδοχείων υφίστανται την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων μέσω της εξωτερικής ανάθεσης και της υπεργολαβίας. Είναι μια πρακτική πολύ συχνή και η οποία εκθέτησε σε κινδύνους ε, το προσωπικό αυτό. Από την Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών, στην οποία εκπροσωπώ την σοσιαλιστική ομάδα, λάβαμε μια, μια πρωτοβουλία για να ε, εκπονήσουμε μια έκθεση όπως αυτή την οποία ε, ζήτησε η Γκούμες της κ. Αλμπιόλ για τα, για τα βήματα οπισθοχώρησης που γίνονται σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων εξαιτία της ε, πολιτικής ε, λιτότητας που έφερε επισφάλεια στην αγορά εργασίας. Πραγματικά ένα πολύ ε, δυσάστο και εξοργιστικό θα έλεγα φαινόμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαντήσει. Την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε αυτός ο περίφημος κοινωνικός πυλώνας. Μπορεί να αποτελέσει μια φετηρία, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο, τίποτα παραπάνω από αυτό. Χρειάζεται να ενισχυθεί με νομοθετικά μέτρα τα οποία θα εγγυώνται την ποιότητα της ε, ζωής ε, των εργαζομένων, γυναικών και ανδρών. Ως σοσιαλιστική ομάδα να σας ενημερώσω ότι ε, προσπαθούμε στις ε, κανόνες ε, τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιλάβουμε και τη, τον, ε, τη σφραγίδα κοινωνικής ποιότητας. Τα ξενοδοχεία, ας πούμε, πέραν των αστεριών που παίρνουν, 4-5 αστεριών και που δείχνουν ότι είναι ένα καλό ξενοδοχείο, θα πρέπει να δούμε πώς συμπεριφέρονται και στους εργαζόμενους, στους εργαζόμενους τους. Οπότε αυτή η σφραγίδα ποιότητας θα μπορούσε επίσης να συμπεριφθεί και στο δικό μας έργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η κυρία Ιστάρα Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τις αναφέρουσες. Εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και να σας πω ότι στην περίπτωση της κυβέρνησης της Ισπανίας έχει ξεκινήσει μια στρογγυλή τράπεζα από τις τελευταίες πληροφορίες που γνωρίζουμε, η οποία ε, σκοπεύει να συζητήσει όλες τις συνθήκες των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ε, οργανώνεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης και από το Υπουργείο Τουρισμού που είναι αρμόδιο για τα θέματα τουρισμού. Συμμετέχουν και πολλές αυτόνομες περιοφέρειες και συμμετέχει και η δική μου των ε, Βαλαρίδων Ίσων και κάποιες άλλες αρκετά τουριστικές αλλά συμμετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή τα βασικά συνδικαλιστικά σωματεία και οι εργοδότες. Ε, από ό,τι γνωρίζω θα συνεδριάσουν σήμερα, ε, ιδίω για να συζητήσουν αρκετά θέματα, αλλά ένα από τα κύρια ζητήματα είναι αυτό το θέμα που θέτετε κι εσείς ε, σήμερα εδώ. Η κυβέρνηση των Βαλερίδων Ίσων, ε, μεταξύ άλλων διεκδικήσεων, ε, η ε, περιοχή είναι τουριστική περιοχή και συζητήθηκε και στο Κοινοβούλιο και ομόφωνα όλα τα πολιτικά κόμματα. Εγώ εκπροσωπώ το Λαϊκό Κόμμα, το Παρτίδο Ποπουλάρ, όπως ξέρετε εμείς είμαστε κυρίως τουριστικά και είμαστε κυρίως Βαλιαρίδες Νήσι και η Φορμεντέρα και εκπροσωπούμε όλες τις ομάδες, ε, λαμβάνουμε υπόψη όλες τις αναφορές που αφορούν τη βελτίωση των εργασιακών συνθήκων, των ωραρίων, την ε, ε, πρόορη ταξιοδότηση, καλύτερο έλεγχο των επιθεωρήσεων εργασίας και όλα αυτά έγιναν δεκτά από την κυβέρνηση των Βαλαιοδονήσεων και θα συζητηθούν εξ ονόματος ε, όλων των βουλευτών ε, στην ε, στρογγυλή αυτή τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Σήμερα ένα από τα σημαντικά νέα από την αυτόνομη περιφέρειά μου έχει μια είδηση που αναφέρεται με τίτλο «Κοινό μέτωπο» για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα πρόορισης ταξιοδότησης και να δεχτούμε όλα τα αιτήματα του Σωματείου Λασκέλης. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι αυτό το βήμα, αυτή η επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε, είναι το κατάλληλο βήμα για να συζητηθούν αυτά τα θέματα και σήμερα έχουμε και τα αιτήματα, έχουμε τους αρμόδιους υπουργούς, τις αρμόδιες αρχές, ε, τους εργοδότες, γιατί φυσικά πρέπει να υπάρξουν και συλλογικές συμβάσεις και τα συνδικαλιστικά σωματεία. Ε, η πρότασή μου λοιπόν είναι είναι να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και να παρακολουθούμε μέχρι να ολοκληρωθούν τα θέματα, διότι είναι καθόλου εύλογο αυτό το ερώτημα, αλλά πρέπει να αποτανθούμε και σε αυτή την επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε και που συνεδριάζει από ό,τι μου λένε ονομάζεται, μισό λεπτό κάπου το έχω σημειώσει, Επιτροπή για την ανάλυση της απασχόλησης στον τομέα ε, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ε, από τις ειδήσει που έχω, σε αυτό το σώμα θα γίνει αύριο η πρώτη συνεδρίαση και η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων θα ε, λάβει υπόψη της και όλα τα αιτήματα των εργαζομένων. Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει αυτή η Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε ε, για να δούμε τι κάνει η κυβέρνηση των Βαλαιαρίδων, η κυβέρνηση της Βαλένθια. Έχουμε ε, αρκετούς ε, και εκεί ε, θα αναφέρουμε και τις ανησυχίες μας και προσυπογράφουμε φυσικά και όλα όσα λέτε κι εσείς. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί μπορούμε πραγματικά σε αυτή την Επιτροπή να κάνουμε τα αιτήματα και έτσι μπορεί να υπάρχει η αλλαγή. Γιατί νομίζω ότι στο Κοινοβούλιο στις Βαλεαρίδες νήσους όλες οι πολιτικές δυνάμεις συμφώνησαν και πιστεύω ότι θα έχουμε ο τέλος, ε, διότι πραγματικά το παρακολουθούμε το θέμα. Ευχαριστώ τη Ρώσα και τώρα να καλωσορίσω την κυρία Γιάλα Σέντερ στην Επιτροπή και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βίκστρομ και ευχαριστώ πάρα πολύ ε, να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου, ε, όπως και οι συνάδελφοι, τις εκπροσώπους ε, του Σωματείου Λασκέλης ε, αυτές τις εργαζόμενες οι οποίες έγινε ένα πολύ σημαντικό αντιπροσωπευτικό κίνημα και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου διότι και η Αυτόνομη Περιφέρεια των Βαλαιαρίδων υποστηρίζει τα μέτρα ε, τα οποία πρότειναν και οι σοσιαλιστές ε, μαζί με το Παρτίδο Ποπουλάρ, το Λαϊκό Κόμμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και καταρχάς θα ήθελα να σας συγχωρώ, διότι αν αύριο είναι η συνεδρίαση και εσείς βρίσκεστε εδώ, σημαίνει ότι σε κάτι χρησιμεύσε όλη αυτή η πορεία που ξεκινήσατε μέχρι τις Βρυξέλλες. Και θα ήθελα να απευθυνθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, όπου γίνονται συστάσεις προς τις κυβερνήσεις των χωρών ανάλογα με την οικονομική, μακροοικονομική κατάσταση, ε, προκύπτει σαφές ότι στην περίπτωση ε, των ε, ε, ξενοδοχείων, όπως είπαν και οι αναφέρουσες, έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάκαμψη και υπάρχουν ωφέλη για τον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αλλά αυτό δεν αντανακλάται ε, και στους μισθούς. Και επειδή υπάρχουν συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, για παράδειγμα στη Γερμανία υπήρχε σαφής ε, ε, σύσταση να αυξηθούν οι μισθοί όταν διαπιστώνεται ότι η οικονομία μιας χώρης, ε, στην Γερμανία μάλιστα έχουμε φτάσει και σε σκανδαλώδη ύψη, αλλά όταν βελτιώνεται η οικονομία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πρώτη η οποία συστήνει στις χώρες ε, να υπάρχει και μια αντιστάθμιση των μισθών με την κατάσταση της εργασίας. Θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατά πόσο η Γενική Διεύθυνση Απασχόληση μαζί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομίας θα μπορούσαν να κάνουν τέτοιες συστάσεις. Διότι αν όντω αναγνωρίζεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ότι η Ισπανική οικονομία έχει πολύ καλά ποσά σε μακροοικονομικά στοιχεία και κυρίως στον τομέα των ξενοδοχείων ε, και πηγαίνει καλύτερα τα τελευταία δύο χρόνια ε, και έχουμε φτάσει και στο 16% αύξηση, θα ήταν δίκαιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει στην, στην Ισπανική Κυβέρνηση να αυξήσει τους μισθούς του συγκεκριμένου κλάδου για να μπορέσει να υπάρχει κατάλληλη αντιστάθμιση και να ε, λαμβάνει υπόψη και τη βελτίωση και τα ωφέλη του κλάδου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κούνεβα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστούμε και τις ε, καμαριέρες από το Κέλλη Έχουμε συνεργαστεί μαζί τους ε, και στην Επιτροπή Απασχόλησης πριν καιρό μαζί με την Τάνε Γκονζάλες. Νομίζω ότι ακολουθώντας τον τρόπο που λειτουργούν οι ομάδες, όπως είπε και η πρόεδρος της Επιτροπής μας, θα πρέπει να προτείνουμε την κατάθεση ερώτησης προς, ε, την Επιτροπή. Τα εργασιακά προβλήματα των εργαζομένων στον ε, τουρισμό δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Ε, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα προβλήματα των εργαζομένων σε αυτό το κλάδο ε, λίγο πιο αναλυτικά και πιο συγκεκριμένα όπως ε, παρακολουθούμε και ρυθμίζουμε την εργασία των εργαζόμενων της μεταφοράς. Αυτός είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πολύ ευάλωτος πολύ δύσκολο να ρυθμιστεί. Και νομίζω ότι πρέπει να, να δούμε πώς θα μπορεί να υπάρχει μια ρύθμιση για τους ξενοδοχοϊπαλληλούς έτσι ώστε να έχουν μια αξιοπρεπής εργασία. Γι' αυτό μίλησα και, και στο σύνοδο, στην στη Κοινωνική Σύνοδο στην Γκέτεμπορκ την προηγούμενη εβδομάδα. Προέταξα τη σημασία των εργασιακών συνθήκων και της αξιοπρεπούς εργασίας και αμοιβής με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό το θέμα δεν είναι μόνο, μεμονωμένο. Πρέπει να δώσουμε ευκαιρία στα συνδικάτα, στους εργαζόμενους να αποφασίζουν τι αμοιβέ να συναποφασίζουν τις αμοιβές τους. Ωστόσο αφήνω ότι συμφωνώ ότι η αναφορά πρέπει να μείνει ανοιχτή και να αξιοποιήσουμε και την πρόταση της κυρίας ε, Εστάρας και φυσικά να μιλήσουμε με τους συντονιστές μας στο τέλος. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ η κυρία Στανόκα. Και σας παρακαλώ να θυμάστε ότι η διερμηνία θα σταματήσει στις 12.30 και θα ήθελα να έχουμε χρόνο να δώσουμε το λόγο ε, και στις αναφέρουσες. Ε, η κυρία Στανόκα, θα είμαι πολύ σύντομη κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αναφέρουσες και θα ήθελα να συμφωνήσω με την πρόταση η αναφορά αυτή να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης, ε, διότι είμαι μέλος του δικτύου ε, ΠΕΤΗ. Νομίζω ότι αυτό θα είναι χρήσιμο. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη με τις ενέργειες της Επιτροπής όσον αφορά την αναφορά αυτή. Δεν νομίζω ότι ήταν επαρκής ε, αντίδραση. Γι' αυτό θα πρέπει η ε, Επιτροπή να βελτιώσει την, ε, τον χειρισμό αυτής της αναφοράς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έτσι έκλεισε ο κατάλογος των ομιλητών και δίνω το λόγο πάλι στην κυρία Μουνιός Ροντρίγες για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Ε... Θα ήθελα να σας ε, πω ότι αντιλαμβανόμαστε πως ε, όλοι μας κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση, έχουμε τις ίδιες διεκδικήσεις. Ε, ε, α, τώρα μας ζητούν να, να εμπιστευτούμε αυτούς που εδώ και, εδώ και τόσα χρόνια από το 2012 καρνούνται τα δικαιώματά μας. Εδώ και πέντε ε, χρόνια ζούμε σε συνθήκες ε, ασθενειών και ε, επισφάλειας ε, και μας ζητούν να συζητήσουμε και να τα βρούμε με αυτούς τους είδους εργοδότες. Δεν υπάρχει καμία, δεν, δεν θέλουμε κανένα καινούριο νόμο. Υπάρχει ο νόμος. Αυτό που ζητούμε απλώς είναι να εφαρμοστεί ο νόμος, να συμμορφωθούν οι εργοδότες με τον νόμο. Και μιλάμε για την υγεία μας. Ε, είναι ένα αμφισβήτητο δικαίωμά μας. Ε, μας ζητούν να συζητήσουμε σε μια επιτροπή εργασίας ε, για τα επόμενα 3, 4, 5 χρόνια και για να λέει εκδοθεί καινούρια νομοθεσία. Υπάρχει νομοθεσία. Μη μας ζητήσετε, να, μη μας ζητάτε να πάμε σε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή για να συζητήσουμε. Εδώ βλέπετε πώς είναι τα χέρια μας. Σας παρακαλώ πολύ μην μας παραπέμψετε κάπου αλλού. Okay. So I think we are ready to take a decision. Νομίζω πως μπορούμε να πάρουμε απόφαση. Προτείνω να κρατήσουμε την αναφορά αυτή ανοιχτή, αυτό είναι σημαντικό, και να δούμε την οδηγία 89391 περί ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στο χώρο και να δούμε να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να εφαρμόζεται σωστά. Οπότε θα ήθελα ως Επιτροπής να στείλουμε μια, μια επιστολή στον Υπουργό Απασχόλησης και να μας εξηγήσει πώς βλέπει αυτή την οδηγία αν θεωρούν ότι έχει εφαρμοστεί πλήρω ή όχι και αν δεν έχει εφαρμοστεί πλήρω να τους ενθαρρύνουν να την εφαρμόσουν. Όπως είπατε και εσείς, η νομοθεσία υπάρχει, το θέμα είναι η εφαρμογή της. Θα ήθελα επίσης να διευρύνουμε λίγο το πεδίο αυτής της επιστολής και να ρωτήσουμε το Υπουργείο τι μέτρα έχει λάβει ή δεν έχει λάβει για να βελτιώσει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. και επίσης να στείλουμε την αναφορά αυτή και στην Επιτροπή Απασχόλησης. Να υπογραμμίσουμε στην επιστολή μας ότι δεν τους λέμε απλώς τι πιστεύουμε, αλλά ότι θέλουμε να απαντήσουν το Υπουργείο, δηλαδή στην Επιτροπή μας, με λεπτομέρειες. Γιατί πιστεύω και γνωρίζω ότι όταν συντάσσουμε αυστηρές επιστολές παίρνουμε πιο ειλικρινείς απαντήσεις. Έτσι έχει η κατάσταση. Και όταν λάβουμε την απάντηση των Ισπανικών αρχών θα πάρουμε απόφαση για το πώς θα συνεχίσουμε. Θα ήθελα επίσης στην επιστολή να υπογραμμίσουμε ότι υφίστανται βέλτιστες πρακτικές ε, τις οποίες ε, έχουν εφαρμόσει άλλα κράτη-μέλη. Αλλά και στην Ισπανία πιστεύω Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η κατάσταση είναι τόσο άσχημη παντού. Κάπου θα υπάρχουν ε, φώτα στο τούνελ, στην άκρη του τούνελ. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και από τα άλλα κράτη-μέλη ενδεχομένω, τα οποία αναζητούν βέλτιστε πρακτικέ. Επίσης ε, θα πρέπει να προσθέσουμε και ένα απόσπασμα για τον κοινωνικό πυλώνα ο οποίος μόλις ε, εγκρίθηκε. Τι σημαίνει κοινωνικός πυλώνας? Σημαίνει ότι στην Ευρώπη πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε όλους τους ανθρώπους σαν να είναι ανθρώπινα όντα. Συμφωνούμε? Βλέπω ότι συμφωνείτε. Ινές? Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και ταυτόχρονα, αν μπορούμε να απαιτήσουμε από την ε, Κομισιόν, μάλλον αναφέρουμε ότι δεν είναι αρκετή η απάντησή της και ζητούμε να επιβεβαιώσουν, να επαληθεύσουν το κατά πόσον η οδηγία εφαρμόζεται από τις Ισπανικές αρχές. Γιατί ε, η Κομισιόν είναι ο θεματοφύλακας ε, το, της ε, νομοθεσίας και πρέπει να μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. ενώ. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαληθεύσει και το κατά πόσον συμμορφώνεται το Ισπανικό κράτος με την οδηγία. Ναι, σύμφωνοι, λέει η Πρόεδρος, ε, Επιτροπή πρόκειται για οδηγία, όχι για κανονισμό αλλά και η οδηγία θα πρέπει να τη χάνει σεβασμού. Και η Κομισιόν πρέπει να παρακολουθεί το κατά πόσον οποιαδήποτε χώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ισπανία, συμμορφώνεται πλήρω με την οδηγία αυτή. Κυρία Γιαλασέντερ, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα το κάνουμε και θα περιμένουμε από την Κομισιόν να είναι πολύ πιο συγκεκριμένη την επόμενη φορά να μας ε, απαντήσει για τον κοινωνικό διάλογο, για το, το διάλογο, για το περιεχόμενό του. Συμφωνώ και με τις δύο προτάσεις, και της Πρόεδρου και της κυρίας Σινέσα Γιάλα. Εγώ επιπλέον θα ήθελα να σας πω το εξή. Το Υπουργείο θα απαντήσει ότι έχει ε, συστήσει ε, μια, ένα συμβούλιο ε, με επτά αυτόνομες περιοχές, η Κανάριες Νήσι, η Βαλένθια, η Ανταλουσία, η Μαδρίτη, η Καστίγια Λεών, η Γαλλικία, η Καταλωνία, όλες, ε, πολλές αυτόνομες περιοχές που ε, διοικούνται ε, από διαφορετικά κόμματα μάλιστα. Το Υπουργείο λοιπόν θα απαντήσει ότι έχει δημιουργήσει ένα συμβούλιο και θα ήθελα να στείλουμε μια επιστολή σε αυτό ακριβώς το συμβούλιο για να βοηθήσουμε. Θα έστελνα λοιπόν και εκεί την επιστολή μας διότι το Υπουργείο θα μας πει έχουμε δημιουργήσει αυτό το συμβούλιο για να εξετάσει το θέμα. Η πρόεδρος του, των ε, Βαλεαρίδων μπορεί να ε, μεταφέρει και τη δική μας άποψη. Ε, εγώ θα έστελνα την επιστολή μας και στο Συμβούλιο αυτό. Ευχαριστώ κυρία Αλμπιόλ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση της Προεδρού να ζητήσουμε πληροφορίες από την Επιτροπή Απασχόλησης και να στείλουμε φυσικά και την επιστολή στο Υπουργείο Απασχόλησης στις Ισπανικές Αρχές ρωτώντας τι έχει γίνει επί του θέματος, τι σκοπεύουν να κάνουν, τι μέτρα έχουν ληφθεί. Ε, προφανώς βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ε, ε, ελέγχει το κατά πόσον τηρείται η οδηγία και πρέπει να αποτανθούμε σε αυτούς. Ε, συμφωνώ και με την πρόταση της κυρίας ε, Εσταράς. Ε, ναι, μεν ε, πολλές φορές δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε όλες τις επιθυμίες των αναφερόντων, έρχονται με πολλά αιτήματα και δεν μπορούμε να τηρήσουμε τα πάντα, αλλά σίγουρα δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι για τα πράγματα τα οποία είπαν ότι δεν θέλουν. Αν είπαν ότι δεν θεωρούν ότι αυτό η Επιτροπή είναι ο χώρος στον οποίο εκπροσωπούνται. Ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε τίποτα ε, για όσα πράγματα δεν ζητούν. Ναι, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλε τι επιθυμίε. Αν ε, πούνε όμω ότι διαφωνούν με κάτι, εγώ θα προτιμούσα να μην το κάνουμε. Νομίζω ότι αρκεί ε, η επιστολή προς, την, το Υπουργείο προ, να αποτανθούμε στην Επιτροπή κλπ. Αλλά κάτι το οποίο δεν τις βρίσκει σύμφωνες νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να γίνει. Αυτή είναι η απόψή μου. Η κυρία Σταράς Φεραγούτ. Φυσικά αυτό έλειπε. Εγώ να πω δηλαδή αύριο στις αρχές των Βαλεαρίδων Ίσων η πρόεδρο που εκπροσωπεί όλα τα κόμματα να μάθει ότι εσεί διαφωνείτε. Να πάει εκεί αύριο εκεί και πάμε όλοι ικανοποιημένοι που θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τι θέσει σα εκεί. Εσεί θεωρείτε λοιπόν ε, ότι πρέπει να πω στην κυβέρνηση των Βαλαρίδων Ίσων ότι αύριο δεν θέλετε να υπερασπιστούν τι θέσει του. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάμε και εκεί. εκτό μικροφώνου τα σχόλια των αναφερόντων. Το μόνο που λέμε είναι ότι ε, να πούμε ότι εμείς ως Επιτροπή Αναφορών θέλουμε να εισακουστούμε. Αν εσείς θεωρείτε όμως ότι η αποστολή φτάνει ε, προς το Υπουργείο, ό,τι θέλετε. Αύριο η Πρόεδρος των Βαλαιαρίδων Ίσων θα κάνει αυτό που κάνετε και εσείς στις Επιτροπές Αναφορές. Ε, δεν ξέρω, εγώ το έκανα για να βοηθήσω. Θα κάνω ό,τι έκαναν μέχρι τώρα. Τίποτα δηλαδή. Πολύ καλά. Ακούστε, η Επιτροπή μου τώρα ξαφνικά γίνεται ένα πεδίο διαμάχης εσωτερικού ισπανικού θέματος μεταξύ γυναικών. Νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε εδώ. Υπάρχει μια πολύ καλή πρόταση για το τι θα κάνουμε και αυτό θα κάνουμε. Και τώρα θα ήθελα να σα δώσω εσάς το λόγο που ταξιδέψατε από πολύ μακριά στις Βρυξέλλες, ε, να φτάσετε στις Βρυξέλλες και ελπίζω να καταφέραμε να εκπληρώσουμε τις ελπίδες και τις επιθυμίες σας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα και θα κάνουμε αυτά που είπα προηγουμένως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις θέσεις μαζί μας και ελπίζω να αφήσετε και ένα από τα μπλουζάκια. Είναι πολύ ωραία και δείχνουν τη δύναμη της, ε, ε, των ανθρώπων, τι μπορούν να κάνουν όταν συνεργάζονται και ενώνουν τις δυνάμεις τους. Ε, κάτι μας διδάξατε εσείς εδώ σήμερα, διότι Νομίζω σήμερα είχα την πιο δύσκολη δουλειά στο Κοινοβούλιο Είχαμε πολύ δύσκολη ψηφοφορία προηγουμένως ε, ε, και όταν βλέπουμε τι γίνεται όταν δεν μπορούν να συνεργαστούν οι άνθρωποι, τσακώνονται, κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν διχασμό ε, και εσεί δείχνετε κάτι διαφορετικό. Πώ μπορούν να ενωθούν οι άνθρωποι και να προσπαθήσουν με αξιοπρέπεια να παρουσιάσουν τι ανάγκε του και τα αιτήματά του και μα διδάξατε πάρα πολλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για το δίδαγμα. καλή επιστροφή σα εύχομαι και να είμαστε σε επαφή. Η αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή. Και σε όλους σε ε, καλή όρεξη. Θα τα πούμε στις 2.30.